Państwa, Κυρίες και κύριοι, ξεκινούμε με μια μικρή καθυστέρηση. Είναι παρόντες νομίζω οι περισσότεροι συνάδελφοι. Δεν είναι συνηθισμένη η ώρα για τη συνάντηση της Επιτροπής μας. Ξέρω ότι υπάρχει μια επικάλυψη με κάποια θέματα στη ημερήσια διάταξη, θα προσπαθήσουμε στο μέλλον να το αποφύγουμε. Λοιπόν, έγκριση ημερήσια διάταξη. Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται. Σας ενημερώνω ότι η συνεδρίαση είναι σε web stream. Δεν έχουμε διερμηνία στα σλοβακικά, μαλτέζικα, εστωνικά και ιρλανδικά. Πριν Πρώτος προχωρήσουμε στην ψηφοφορία για το σημείο 3 και δώσω το λόγο στον κύριο Γιάρα. Θα ήθελα να σας ενημερώσω. Μας το είπε στο ξεκίνημα ο πρόεδρος Σούλτς ότι χθε ο κύριος Μπονάνο, συνάδελφος, σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό ατύχημα. Είχε συνεργαστεί με την Επιτροπή μας Έχουμε κάποιες πληροφορίες για τα... τον αποθανόντα συνάδελφο, για όσοι δεν τον ξέρετε. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να κρατήσουμε ενό λεπτού συγγύη. tak nieznane są losy ludzkie. Proszę Państwa, zgodnie z zapowiedzią... Αυτά. Τώρα, όπως σας αναγγείλαμε, θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Γιάρ που είναι εδώ. Η κυρία Σέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να καταγραφεί η δυσαρέσκειά μου. Η συνάντηση αυτή συμπίπτει με μια συζήτηση στην Ολομέλεια για θέματα γεωργίας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ε, καταλήξαμε στην κατάσταση αυτή. Να χρειάζεται εν τέλει να αποφασίσουμε αν θα πάμε στην Επιτροπή Γεωργίας ή αν θα μετάσχουμε ή θα παραστούμε τουλάχιστον στην συζήτηση που γίνεται στην Ολομέλεια ταυτόχρονα. Θα παρακαλούσα να το λάβετε υπόψη αυτό και να μην επαναληφθούν παρόμοιες καταστάσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Το είπα και στο ξεκίνημα της ε, παρέμβασής μου. Θα προσπαθήσουμε στο μέλλον να αποφύγουμε καταστάσεις όπως αυτές. Προφανώς ε, όμως ε, υπάρχουν κάποια τεχνικά, τεχνικές υποχρεώσεις και μας το επιβάλλουν. Τέλος πάντων θα φροντίσουμε, θα προσπαθήσουμε να μην ξαναγίνει. Κύριε Γιά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τρεις παρατηρήσεις. Καταρχάς ε, να ευχαριστήσω, να ζητήσω συγγνώμη και να κάνω μια ανακοίνωση. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της Επιτροπής και κυρίως τους σκιώδεις εισηγητές. Είχαμε τρεις συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών. Και σε κάθε τέτοια συνάντηση ε, ε, έγινα πιο σοφός. Σας ευχαριστώ για την επικοδομητική συνεργασία. Ζητώ συγγνώμη. Σχετικά με την ε, οδηγία για τον προϋπολογισμό. Αποφασίσαμε ότι εάν ε, έχει ο τομέα ε, τη γεωργία ε, περισσότερα καθήκοντα, περισσότερε αρμοδιότητε, θα πρέπει να λάβει και περισσότερου πόρου. Λάβαμε πολλέ τροπολογίε που ήταν πολύ ενδιαφέρουσε ω προ το περιεχόμενο, αλλά στη συνάντηση των σκιωδών είπαμε ότι θέλουμε να, να παραμείνουμε εντός θέματος. Θέλω λοιπόν ε, να παρακαλέσω τους συναδέλφους, των οποίων δεν έχει οθετηθεί η τροπολογία, να θυμούνται ότι κατά τη διάρκεια του ε, ελέγχου ε, της Γεωργίας θα, θα θυγούν τα θέματα αυτά. Και τέλος, μια ανακοίνωση ανακοίνωση, τροπολογία για την παράγραφο 10, προφορική έχουμε και επίσης μία προφορική τροπολογία για την 131 και οι δύο προφορικές τροπολογίες ε, πρέπει ήδη να βρίσκονται στον κατάλογο της ψηφοφορίας. Όταν φτάσουμε στο σημείο αυτό ε, θα πάρω το λόγο, αλλά νομίζω ότι βρίσκονται ήδη στο έγγραφο. Σε ευχαριστώ όλους για την επικοδομητική συνεργασία και που μπορούμε ε, εντός της ε, προθεσμίας ε, να υιοθετήσουμε την έκθεση. Επίσης έχουμε 7 συμβαστικές τροπολογίες, να θυμηθώ να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θα κρατήσουμε τις ευχαριστίες για το τέλος της συνεδρίασης προς εσάς κύριε συνάδελφε. Είναι εξαιρετικά επίκαιρο το κείμενο που συζητούμε και αυτή θα είναι η γραμμή που θα κρατήσουμε μέχρι το τέλος των εργασιών μας σχετικά, που, μόνο το που ξεκινάνε μόνο τώρα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για τις προφορικές τροφολογίες, αλλά προχωρούμε στην ψηφοφορία. Θα προσπαθήσω να το κάνουμε με αποτελεσματικό τρόπο. Τροπολογία 1. υπέρ Χάζακαμπ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 2 υπέρ εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ ευχαριστώ εγκρίνεται τροπολογία 4 υπέρ εγκρίνεται τροπολογία 5 κατά τμήματα Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική α με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχουμε έναν έξτρα από την Άλντε. Βγάλετε μια κάρτα από την Άλντε. Πέρας ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 19 υπέρ εγκρίνεται. 20 Προπολογία 20 καταπίπτει, 21 καπούτο υπέρ εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά απορρίπτεται. 23 υπέρ, εγκρίνεται. 24 υπέρ, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά απορρίπτεται 31 υπέρ κατά απορρίπτεται 32 υπέρ κατά απορρίπτεται 33 υπέρ εγκρίνεται 34 υπέρ εγκρίνεται 35 υπέρ Κατά. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 40 Ζητήθηκε έλεγχος για την 39. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 39. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 49. Συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. 40. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 54 υπέρ κατά απορρίπτεται. Η τροπολογία 55 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Ευχαριστώ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 58 άρχεται η ψηφοφορία. της ψηφοφορίας. Έχετε δίκιο, εγκρίνεται. 59 έχει αποσυρθεί 60 υπέρ κατά θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 60 και η ίδια πλειοψηφία είναι αρχίζει η ψηφοφορία για την 60 ευχαριστώ πολύ Ας ψηφίσουμε κανονικά. Επαναλαμβάνεται. Απορρίπτεται. Ευχαριστώ. Συμβιβαστική C. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 67 τροπολογία υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Μια προφορική τροπολογία στην παράγραφο 10 της κυρίας Αγγιλέρα. Εντάχει. Στην έκθεση και το είχα πει του εισηγητή είχαμε κάνει μια ειδική ε, ρήτρα διαφύλαξη την κατηγορία 2, αλλά στην κατηγορία 3 με τίτλο Ασφάλεια και πολίτες περιλαμβάνεται ό,τι έχει να κάνει με μέτρα για την υγιεινή των ζώων και των φυτών, το φυτογενομικά. Και εδώ θα έπρεπε στην τροπολογία αυτή να υπογραμμίσουμε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πόροι. το θέμα της προστασίας των πόρων η τροπολογία λοιπόν λέει, εκφράζει τη λύπη της ότι τα υπόλοιπα που απευθύνονται σε φυτογενομικά μέτρα βρίσκονται στην κατηγορία 3 του παρόντος ε, πολιτούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου και υπογραμμίσει ότι οποιαδήποτε μείωση ή αναδιανομή αυτής της γραμμής του προπολογισμού θα προϋποθέτει μια απειλή για την ε, ασφάλεια των τροφίμων και τη υγιεινή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην υπάρχουν λιγότεροι υπόλοιποι δηλαδή, στην κατηγορία 3 για την υγιεινή ζώων και φυτών από ό,τι τώρα. Επειδή δεν βρίσκεται στην κατηγορία 2 θα μπορούσε να ξεχαστεί αυτό. Ευχαριστώ. Ζήτησαν υπάρχουν αντιρρήσει να μου πει κάποιο. Ποιοι είναι υπέρ τη τροπολογία αυτής, τη προφορική τροπολογία. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική D. Άρχεται η ψηφοφορία. Το τμήμα 1 είναι γιατί είναι κατά τμήματα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας Ευχαριστώ, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα της συμβιβαστικής D, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται και αυτό. των υστέρων δεν γίνεται. Όχι. Δεν ήταν σαφές αν έχουμε ήδη ψηφίσει το δεύτερο τμήμα ή αν είμαστε ήδη στην 77. Δεν ήταν σαφές. Παρακαλώ να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Κύριε συνάδελφε, έξυπνη ερώτηση. Αυτό ήταν ηλεκτρονική η ψηφοφορία, ήταν ηλεκτρονική. Ψηφίσαμε το κείμενο, δεν αλλάζει, προχωρούμε. το απολογεί 77, λέει ο πρόεδρος, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 78 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος. Τροπολογία 79. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 80 υπέρ. Εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 83 υπέρ. Εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 87 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 91 υπέρ κατά απορρίπτεται 86 Ας γίνει έλεγχος για την ηλεκτρονική έλεγχο 91 άρχεται η ψηφοφορία 91 Ευχαριστώ πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται Μικρή ψηφοφορία, αλλά πρέπει. 86 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο. Ηλεκτρονικό έλεγχος για την 88. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 90 υπέρ. Εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά. Απο, απορρίπτεται. Συμβαστική ή e με ηλεκτρονική, ε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορια Ευχαριστώ. Τροπολογία 101. Υπέρ. Απορρίπτεται. 103. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική F. Υπέρ. Ε, ηλεκτρονικά η συμβαστική F. Συγγνώμη. Άρχεται η ψηφοφορία για την συμβαστική F. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 114 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική G. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 125. Υπέρ. 125 κατά. Απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 128 υπέρ. Διορθώνει ο πρόεδρος. 127 ταραμπέλα. Συγγνώμη κύριε ταραμπέλα. Υπέρ τη 127 εγκρίνεται. Ήξερα ότι θα εγκρινόταν, γι' αυτό δεν την πρότεινα. 128 άγνιο υπέρ εγκρίνεται. 129 υπέρ εγκρίνεται. 140 υπέρ κατά απορρίπτεται. Έλεγχος για την 130. Άρχεται η ψηφοφορία. της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία από τον πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών, ο κ. Σαχτουή. Είναι μια προσωπική τροπολογία που υπογραμμίζει πόσο ενδιαφέρον θα ήταν να υπάρξει ένα ασφαλιστικό ταμείο που θα επιτρέπει σε περίοδους ε, μεγάλης αυξομοίωσης των τιμών όταν πέφτουν οι τιμές και θέλουμε να θρύνουμε τους παραγωγούς να μειώνουν το όγκο παραγωγής, να τους πείθουμε ότι θα έχει κάτι θετικό η μείωση της παραγωγής τους για να ξαναβρούμε την, ξαναβρούμε την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και να επιτρέψουμε την άνοδο των τιμών. Αυτή είναι η προφορική τροπολογία που αλλάζει την αρχική 131. Ευχαριστώ. Ήταν υπουργό οικονομικών στην γαλλική κυβέρνηση και εκτιμούμε την τροπολογία του. Για το πρώτο τμήμα, υπέρ Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Εγκρίνεται η τροπολογία. Τελική ψηφοφορία. Το με τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν θα γίνει ηλεκτρονικά. Γνωμοδότηση για άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ για την γνωμοδότηση και τις τροπολογίες. Μήπως θα ήθελε να πει κάτι ο εισηγητής. Όχι. Ο κύριος Ιάρ, Κύριε Πρόεδρε, ήταν πολύ καλή δουλειά που κάναμε και ήμασταν ε, ενωμένοι όσον αφορά τις αποφάσεις. Τώρα θα πρέπει να πείσουμε τους συναδέλφους από την Επιτροπή Προϋπολογισμού ε, για την σωστή μας αυτή άποψη. Αν το πετύχουμε, αυτό θα είναι μια προσπάθεια οικοδόμησης εμπιστοσύνη, όχι μόνο για την γεωργική πολιτική της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη ε, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Είναι σημαντικό όσον αφορά τον προπολογισμό μας να σταθούμε στο πλευρό των γεωργών μας. Κυρίες και κύριοι, το βλέπω σε πολλές συνεδριάσεις η Επιτροπή Προϋπολογισμού να είναι υπέρ κάποιων από τις ιδέες μας, αλλά πρέπει να πείσουμε και τους συναδέρφους και από άλλες επιτροπές. Ε, φτάνουμε στο επόμενο θέμα της ε, ημερησίας διάταξης. Ε, η συγκητής είναι πάλι ο κύριος Γιάρ. Προϋπολογισμός 2017. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω τους και τις εισηγητές. Ε, είχαμε ε, και πάλι είχαμε 48 ε, τροπολογίες. Έχουμε εκπονήσει τρεις συμβαστικές τροπολογίες. Και θα πρέπει όσον αφορά τον προϋπολογισμό και την γεωργική πολιτική να δουλεύουμε πολύ σωστά, διότι το 2017 πετύχαμε αυτά που θέλουμε, αλλά το 2017 είχαμε υποσχεθεί στους γεωργίους μας να διαθέσουμε τους πόρους που χρειάζονται. Εάν δούμε να αυξάνονται οι τιμές και οι γεωργοί να έχουν ένα ε, καλό εισόδημα, τότε θα έχουμε πετύχει το στόχο μας. Και ελπίζουμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στην επίταξη του στόχου αυτού με την ε, σημερινή έκθεση. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, προχωράμε στην ψηφοφορία. Συμβιβαστική τροπολογία Α, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Ζητώ συγγνώμη. Συμβιβαστική τροπολογία Β, διορθώνει ο Πρόεδρος. Συμβιβαστική Β, αρχή τη ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 13. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Ε, η ηλεκτρονική επαλήθευση. Εντάξει, ε, ελέγχουμε την 14, αρχή της ψηφοφορίας, τροπολογία 14 επαλήθευση. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Με μικρή πλειοψηφία. 15 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική C, γάμα. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική D, δέλτα, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση 34 αρχή της ψηφοφορίας λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται 35 υπέρ κατά απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά απορρίπτεται. 36 υπέρ εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση αρχή της ψηφοφορίας για την 38. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική ε. Αρχή της ψηφοφορίας για τη συμβαστική ε. Λήξη της ψηφοφορίας. εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ πολύ. Η γνωμοδότηση για τον προϋπολογισμό 2017 εγκρίθηκε. Συγχαίρω όσους συμμετείχαν. Θέλει να προσθέσει κάτι ο κ. Όχι. Και εγώ είδα την ικανοποίησή του. Ο κύριος Σεγιάρη. η καλή συνεργασία μου ανοίγει την όρεξη για περισσότερη συνεργασία. Ευχαριστώ και πάλι όλους τους συναδέρφους και τους σκιώδεις εισηγητές. Ελπίζω να μας πείτε το ίδιο και στο τέλος της εργασίας που θα έχουμε ολοκληρώσει για τον προϋπολογισμό. Όταν εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό για το 2017 στην τελική του μορφή. Περνάμε στην έκθεση της εισηγήτριας Εστέρ Έρανθ Γκαρθία, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Είναι μια έκθεση γνωμοδότησης, την οποία υποβάλλουμε στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις τροπολογίες, για τις προτάσεις τους, για την επικοδομητική και γενναιότερη στάση που έχουν επιδείξει όλους τους συναδέλφους από όλες τις πολιτικές ομάδες. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και τη δέσμευση που αναλαμβάνετε. Οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε η έκθεση επί της ουσίας ε, της ε, συναδέλφου να συμπεριλάβει τις προτάσεις μας. Οι έξι συμβιβαστικές τροπολογίες ε, νομίζω συνοψίζουν την άποψη της Επιτροπή μας για αυτό το θέμα. Να σας πω ότι η τροπολογία 108 έχει αποσυρθεί. Ας ξεκινήσει η ψηφοφορία λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε λοιπόν. Να σας πω ότι ορισμένες επιτροπές απορρίπτουν πλήρως και δεν γνωρίζω γιατί συμβαίνει αυτό των, ε, απορρίπτουν τις γνωμοδοτήσεις των επιτροπών που υποβάλλουν γνωμοδότηση. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Εγώ χαίρομαι όταν άλλες επιτροπές ε, συντάσσουν γνωμοδοτήσεις για δικές μας εκθέσεις και πάντοτε τις λαμβάνω υπόψη μου και τις μελετώ προσεκτικά το να λαμβάνει κανείς υπόψη του τους άλλους και το τι κάνουν οι άλλοι δεν αποδυναμώνει τη θέση του, αντιθέτως την ενισχύει κατά τη γνώμη μου και θα πρέπει να κάνουμε τα δέοντα έτσι ώστε η δική μας γνωμοδότηση να συμπεριληφθεί στην έκθεση επί της ουσίας. Άλλωστε η κοινή γεωργική πολιτική συνδέεται άρρηκτα με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τρίτες χώρες. Υπάρχουν εμπορικές ε, συμφωνίες που διαδραματίζουν σήμερα καθοριστικό ρόλο γιατί η αγορά σήμερα είναι παγκόσμια και αυτό έχει αντίκτυπο στην Ευρώπη, στην κοινή γεωργική πολιτική και κατά τη γνώμη μου οφείλουμε όλοι να πράξουμε τα δέοντα έτσι ώστε να αλλάξουν τα πράγματα και να λαμβάνεται υπόψη η άποψή μας και στις άλλες επιτροπές. Λυπούμε που σας κούρασα, αλλά έπρεπε να κάνω αυτό το σχόλιο. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική υπαριθμών 1. Πέρας της ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Με παρατήρηση, με σχόλιο. Η τελευταία πρόταση τη βλέπετε υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 5 υπέρ, εγκρίνεται. 19 υπέρ, εγκρίνεται. 24 υπέρ, εγκρίνεται. 25 υπέρ, εγκρίνεται. 26 υπέρ, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 31 υπέρ, εγκρίνεται. 34 υπέρ, εγκρίνεται. 18 υπέρ, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Νομίζω ότι απορρίβεται, αλλά δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε την 33, παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. με μικρή διαφορά. Συμβαστική 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Η κυρία εισηγήτρια, νομίζω ότι το ίδιο πρόβλημα υπάρχει εδώ, διότι ε, υπάρχει διακοπή στη διερμηνία. Ξαφνικά ε, σταματάει η σύνδεση και δεν ακούμε τίποτα στα ακουστικά μας. Νομίζω ότι και άλλοι συνάδελφοι έχουν αυτό το πρόβλημα. Σβήνεται, δεν ξέρω γιατί σβήνεται. Τώρα σας ακούω μια χαρά, λέει ο Μιλίτρε Και ο κύριος Έρδος, ίσως είναι το μπλοκ εδώ που καθόμαστε. Το ίδιο πρόβλημα έχει και ο διπλανός μου. Σβήνει το μηχάνημα. Ίσως πρέπει να αλλάξουμε θέση. Σβήνει το μηχάνημα. Και σε σένα συμβαίνει, έτσι δεν είναι, ναι. Γνέφει καταφατικά ο διπλανός μου. Να αλλάξουμε θέση. Πράγματι, Ίσως πρέπει πραγματικά να αλλάξετε θέση και αν επαναληφθεί το πρόβλημα να μας το πείτε. 43 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 50 υπέρ. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Ε, εγκρίνεται. είχε καταπίσει, γιατί είχε, είχε καταπέσει, γιατί είχε εγκριθεί το ίδιο. Το ίδιο ισχύει για το 113, πάμε στην 52 υπέρ κατά. Απορρίπτεται. 55 υπέρ. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. 71 της κυρίας Ένθα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 73 υπέρ εγκρίνεται. 74 υπέρ εγκρίνεται. 36 Συμβιβαστική 4 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ομοφόνος. 90 υπέρ. Εγκρίνεται. 92 υπέρ. Εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 97 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 99. Υπέρ. Εγκρίνεται. Η 108 και όπως σας είπα. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 118 υπέρ. Εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται νομίζω, αλλά θα το επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε την 123 ηλεκτρονικά. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με ελάχιστη διαφορά Ψήφα. Εγκρίνεται λοιπόν συγχαρητήρια στον κύριο Μποβέ. 124 υπέρ εγκρίνεται. 125 υπέρ εγκρίνεται. 126 υπέρ εγκρίνεται. 127 υπέρ εγκρίνεται. 128 υπέρ εγκρίνεται. 131 υπέρ. Θέλετε να επαληθεύσουμε. 131 του κυρίου Μποβέ, υπέρ, κατά. Θα το επαληθεύσουμε γιατί νομίζω ότι απερίπτεται. Ψηφίζουμε την 131 του κυρίου Μποβέ, ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 132 υπέρ. Εγκρίνεται. 115 έχει καταπέσει 133 υπέρ εγκρίνεται 134 υπέρ κατά απορρίπτεται 135 της εισηγήτριας υπέρ εγκρίνεται 23 όχι 21 όχι Ψηφίζουμε λοιπόν το σύνολο του κειμένου. Ξεκινάει η ψηφοφορία για το ψήφισμά μας, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Κυρία Ισηγήτρια, σας ευχαριστώ πολύ για την ψηφοφορία. Πολύ ευχαριστώ τους συναδέλφους για το επικοδικό δομητικό τους πνεύμα, για την εργασία τους και ελπίζουμε ότι η Ισηγήτρια από το EFTD, η κυρία Μπεγίν, θα λάβει υπόψη της στη δική μας ε, νομοδότηση. Θα το προσπαθήσουμε πάντως εμείς. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Περνάμε τώρα στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για ένα πρόβλημα επί της ουσίας. Ουσιαστικό. Η αστάθεια των τιμών στην ε, αγορά αγροτικών προϊόντων στις γεωργικές αγορές. Η συγγήτρια είναι η κυρία Ντελαέ. Και θα της δώσω το λόγο για να μας παρουσιάσει ε, το κείμενο αυτό. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι που είστε εδώ παρόντες και παρούσες και αγαπητοί σκιώδεις εισηγητές, θα σας πω κάποια πράγματα που πλαισιώνουν αυτό το θέμα. Πράγματι, η αστάθεια των τιμών είναι ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ και καιρό. Πόσο μάλλον σε αυτή την περίοδο κρίσης, όπου δυστυχώς κανένας κλάδος ε, της ε, γεωργίας ε, δεν βρίσκεται στο απειρόβλητο. Μιλήσατε για τις εμπορικές συμφωνίες και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε επίσης και για τη διπλωματική πολιτική έναντι των τρίτων χωρών και το ρωσικό εμπάργο το οποίο υφίστανται οι Ευρωπαίοι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων. Πληττόμαστε λοιπόν και ε, καλούμαστε ως Ευρωπαίοι να ε, κομίσουμε λύσεις συγκεκριμένες και αυτές. Και όλα αυτά μάλιστα στο πλαίσιο της ανανέωσης και αναθεώρησης της κοινή γεωργικής πολιτικής. Εδώ και αρκετές εβδομάδες δούλεψα με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, με άλλους συναδέλφους βουλευτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να καταλήξουμε σε αυτή την πρόταση και για να καταλάβουμε καλύτερα τα διακυβεύματα που ε, εγείρονται από την αστάθεια των ε, τιμών. Οργανώσαμε διάφορες εκδηλώσεις και θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας, ε, στη διάσκεψη που έγινε παρουσία του καθηγητή Σαλμάν, ειδικού των διεθνών αγορών και γεωργικών θεμάτων πριν από ένα μήνα εδώ στο Στρασβούργο. Είχαμε την ευκαιρία να έχουμε σωστή πανεπιστημιακή και ακαδημαϊκή τεκμηρίωση πίσω από όλα αυτά τα θέματα. Σε λίγες μέρες στο, στο Στρασβούργο οργανώνω και ένα άλλο συνέδριο παρουσία άλλων εμπειρογνωμόνων μεταξύ άλλων και στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην στέλεχος του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας. Και περιμένω να έρθετε, να προσέλθετε, να είστε πολυάριθμοι, πολλοί, όπως και τον περασμένο μήνα. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να σας δώσω κάποια ε, γενικότερα στοιχεία. Στόχος της έκθεσης είναι να διαπιστώσει ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή ως προς την αστάθεια των τιμών και να καθορίσει μακροπρόθεσμους στόχους διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί και για να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα θα ασχοληθούμε στην έκθεση αυτή μόνο με την αστάθεια των τιμών και όχι με τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των κρίσεων ή το επίπεδο ε, της χαμηλότερης τιμής και της διαμόρφωσης της τιμής στην αγορά. Οι τρεις προτάσεις που προβάλλονται στην έκθεση αυτή είναι η διάρθρωση των κλάδων και η συμβασιοποίηση με τις οργανώσεις παραγωγών, η θέσπιση εργαλείων διαχείρισης κινδύνου όπως είναι ε, η ασφάλιση και τα αμοιβαία κεφάλαια και διάφορα ε, χρηματοπιστωτικά εργαλεία για να υπάρχει ε, καλύτερη εξασφάλιση των αγροτών και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε ε, και στο G20 έχει, έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Θέλουμε η έκθεση αυτή να είναι ένα σαφές μήνυμα το οποίο να στέλνεται στους Ευρωπαίους αγρότες για να τους αποδείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι εχθρός τους, όπως πολλοί μπορεί ενδεχομένως να νομίζουν, αλλά ότι επιθυμούμε να τους βοηθήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο. Και ε, περιμένω ε, τις ε, ε, τροπολογίες σας και θα ήθελα αυτό το κείμενο να, καταλήξει, να, να είναι όσο τον πιο ποιοτικό με τη δική σας συνεισφορά. Να μην, να μην ξεχάσω να σας πω Να σας πω ότι τον επόμενο Ιούνιο μέσα ότι στις ο 8 Ιουνίου θα έχουμε συζήτηση και για το Farm Bill και για διάφορα θέματα. 13 Ιουνίου είναι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Ελπίζουμε να το συζητήσουμε στο, στις 8 Νοεμβρίου στην Επιτροπή και να ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Και ελπίζω να ήμουν σύντομη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ για την ε, εισαγωγή σας. Θα ήταν χρήσιμο αν οι σκέψεις σας συμπεριλαμβάνονται στις εργασίε που διεξάγονται αυτή τη στιγμή για την αντιμετώπιση της ε, αστάθειας των τιμών στην παγκόσμια αγορά και στην ενδιάμεση αναθεώρηση ενδεχομένω. Ο κύριος Καπούτο έχει ζητήσει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχά την εισηγήτρια και λέει για την έκθεσή της. Ε, έκθεση σημαντική προφανώς που όπως ε, είπε και η ίδια περιμένει ακόμα την συμβολή των συναδέλφων για τη βελτίωσή τους. Στη φάση αυτή ε, θα προσπαθήσουμε, στη φάση των τροπολογιών θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ή να συμπεριλάβουμε και άλλα θέματα. Εγώ θα σταθώ σε τρία κύριο σημεία. Πρώτον, ανάπτυξη των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου, ιδίω των διάφορων μορφών ασφάλισης και ε, ταμείων αμοιβαία συνδρομής. Νομίζω ότι αυτός ο δεύτερος τρόπος είναι βασικός για να, το Ταμείο Λοβοήθειας Δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να επεκταθεί στην ε, έκθεση. Χρειαζόμαστε Ταμείο Λοβοήθειας στην Ένωση για να παράσχουμε στους γεωργούς μια πραγματική προστασία από τις απώλειες εισοδήματο. Θα πρέπει να υπάρχει ευρύτερη κάλυψη σε, σε σχέση με τα παραδοσιακά μέτρα που λαμβάνουν υπόψη και τα φαινόμενα που με κάποιο τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τον τζίρο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μεταξύ αυτών και οι κίνδυνοι της πορείας της αγοράς. Το Incal Stabilization Tool από αυτή την άποψη που δοκιμάστηκε με επιτυχία και στην Ιταλία και στο Βέλγιο μπορεί κατά την άποψή μου να αποτελέσει μια ουσιαστική καινοτομία στην ευρωπαϊκή προσφορά πολιτικών υποστήριξης σταθερότητας των ε, γεωργικών εισοδημάτων, διότι είναι το μόνο εργαλείο, η μόνη μέθοδος που εξασφαλίζει την διαχείριση κινδύνου από την, το ευμετάβλητο των τιμών. Το δεύτερο θέμα που θέλω να σχολιάσω αφορά στις ε, αντικυκλικές ενισχύσεις. Η συγγήτρια και εμένα, όπως είπε, αποφάσισε να μην προτείνει τέτοια μέτρα είναι μια απόφαση κάπως έτσι τραβηγμένη κατά την απόψή μου. Γιατί σε ένα πλαίσιο μεγάλης αβεβαιότητας ε, για το μέλλον των γεωργικών τιμών που είναι και ασταθείς και χαμηλές, η Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη δράση στις αγορές με την δημιουργία δικτύων ασφάλισης και συστημάτων πρόληψης και διαχείρισης των κρίσεων που πρέπει να στηρίζονται κυρίως σε αντικυκλικές ενισχύσεις που επιτρέπουν στους γεωργούς να έχουν ε, τιμές που να είναι ανταγωνιστικές για αυτούς. Να σημειώσω εν τέλει ότι μικρή μνήα γίνεται σε καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Είχα μιλήσει και με τον επίτροπο κύριο Χόγκαν στο παρελθόν για το θέμα αυτό. Γίνεται μικρή αναφορά, για παράδειγμα, στην εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ούτε αναφέρεται στην έκθεση. Αντίθετα, νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε και να υπογραμμίσουμε το ρόλο αυτό, ε, τον ρόλο του οργάνου αυτού και τις παρεμβάσεις του για να μπορέσουμε να έχουμε ευκολότερα στη διάθεσή μας εργαλεία κατά αντικυκλικά που θα βοηθήσουν τους γεωργούς και μπορεί να αντιμετωπίσει ή άλλα μέσα που μπορεί να τη χρησιμοποιηθούν ως αντικυκλικά μέσα. Προφανώς στις επόμενες εβδομάδες θα ε, προτείνουμε κείμενα για να έχουμε και θα ζητήσουμε για να υπάρξουν ε, από κοινού λύσεις. Εκτός στο μικροφόνο πρόεδρος. Είναι γεγονό ότι οι πολλοί παράγοντε επηρεάζουν την αστάθη, τις τιμές, τη σταθερότητα των τιμών. Δεν μπορούμε όμω σε μια έκθεση να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Γιατί το πρόβλημα είναι πολύ σύνθετο. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σας. Καταλαβαίνω ωστόσο και την πρόθεση της εισηγήτριας να μην προσπαθήσει να καλύψει τα πάντα. Κύριε Σράγερ, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση αυτή συνδέεται με το θέμα που συζητιέται αυτή τη στιγμή στην Ολομέλεια. Ιδιαίτερα χαίρομαι με αυτά που έχει καταγράψει εδώ η Αντζελίκ. Θα ήθελα όμως να μου πει τι πιστεύει για τον νόμο πλαίσιο για, την, για τον ανταγωνισμό, διότι πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε νομοθετική βάση για όλα αυτά. Και το λέω αυτό διότι στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο συζητήσαμε το πρόβλημα των τιμών και το τελικό αποτέλεσμα ήταν ότι δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία. Εάν δεν υπάρχει νομοθεσία, είναι δύσκολο να πετύχει ο σε μια λογική τιμή για τα προϊόντα του. Όσον αφορά τις οργανώσεις των παραγωγών. Και αυτό το θέμα συνδέεται με τους συνεταιρισμούς. Ο διευθυντής κοιτάει να δει τι κέρδος υπάρχει και τα δύο τρίτα της τιμής ε, έχουν να κάνουν με την μεταποίηση, ενώ μόνο το ένα τρίτο καταλήγει στον γεωργό. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν ε, οι γεωργοί να έχουν σωστές τιμές για τα προϊόντα τους. Ε, και θέλω να μιλήσω και για το μποϊκοτάς της Ρωσίας. Η Κομισιόν δεν κάνει κάτι εδώ, ίσως θα πρέπει εμείς να κάνουμε κάτι τα πιστοποιητικά εξαγωγών θα μπορούσαν να αποτελέσουν λύση. Ξέρω ότι πολλοί είναι κατά αυτού. Νομίζω όμως ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε πολλά με τον τρόπο αυτόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μασάου. Euh, Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ε, του 12 οδήγησε την γεωργία στη Γαλλία σε μια κατάρρευση. Έχουμε συγκέντρωση, μείωση των εκμεταλλεύσεων, υπερχρέωση, πτωχεύσεις. Πρέπει να σταματήσουμε πλέον να εξατόμεθα επισυριστικά και να ενισχύσουμε τις εξαγωγές. Επίσης, να αποκτήσουμε εκ νέου την επισητιστική κυριαρχία και να ε, περιορίσουμε το ελεύθερο εμπόριο. Αυτό είναι κάτι που ελπίζω. Με εξέπληξαν τα λόγια της συναδέλφου κύριε Ντελαέ. Ομολογώ ότι εξεπλάγιν που διάβασε ότι ένα κείμενο που η ψεύτικη δεξιά, όπως είναι η κυρία Ντελαέ, υποστηρίζει τις αρνητικές, αναφέρει τις αρνητικές συνέπειες της ΚΑΡΤ, της γεωργικής πολιτικής, που την έφτιαξε και υποστηρίζει την ταύτα, την ε, απελευθέρωση του, της γεωργίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Υποστηρίξατε και τις διεθνείς συνθήκες μεταξύ αυτών με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, η διαπραγμάτευση των οποίων ξεκίνησε και που θα συντρίψει περαιτέρω την κατάσταση των Ευρωπαίων Γεωργών. Η αστάθεια των τιμών είναι στο DNA των φιλελεύθερων. Αν δεν θέλετε αστάθεια, πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω από ένα παρατηρητήριο, να βγούμε από την κουλτούρα της κερδοσκοπίας και να εξασφαλίσουμε ελάχιστες τιμές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, η απελευθέρωση των τιμών των γεωργικών προϊόντων με, ε, με την αποσύζευξη τελικά έχουν πλήξει την γεωργική παραγωγή η οποία υφίσταται κερδοσκοπικές πιέσεις προς τα πάνω και προς τα κάτω. Η κυρία Ντουελαέ μίλησε για τις πρώτες ύλες, όμως εγώ θεωρώ ότι ο εισηγητής αυτό που λέει είναι ότι είναι ανησυχητικέ οι τιμέ των πρώτων υλών και οι χαμηλέ αυτέ τιμέ θα μπορούσαν να κρατήσουν για 10 χρόνια και δεν πρόκειται να βελτιωθούν. Άρα δεν είναι περαστική η κρίση αυτή, είμαστε στο τέλος ενός ανωδικού κύκλου και το κείμενό σας δεν κάνει τίποτα για να βελτιώσει την κατάσταση της γεωργίας μας. Το μόνο που κάνει είναι να ε, φτωχαίνει ακόμα περισσότερο τους αγρότες και υπάρχουν χώρες που αξιοποιούν την κρίση για να κερδίσουν όλο και περισσότερα χρήματα. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συντάξουμε μια έκθεση για να δείξουμε ότι πράγματι υπάρχουν εργαλεία και μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση των αγροτών μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Αντρία, αλλά παρακαλώ όχι τέτοιες αντιθέσεις έντονες. Σας ευχαριστώ. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα και το είπατε και εσείς στην εισαγωγική σας παρατήρηση κύριε Πρόεδρε και η κυρία Ντουελαέ το, το παραδέχθηκε. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω για τη δουλειά της, για τη μέθοδο που χρησιμοποίησε Σε αυτό το τομέα, ξέρετε, η αλήθεια δεν είναι εύκολη και πρέπει να εργαστούμε συλλογικά. Και στα συνέδρια που διοργάνωσε φάνηκε αυτό. Είναι καλό που έχουμε ένα πρώτο κείμενο και μπορούμε να στηριχθούμε πάνω σε αυτό και να το λάβουμε υπόψη μας για την επόμενη μεταρρύθμιση. Δύο γενικές παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Οι προτάσεις σας Πράγματι απαντούν, αλλά μόνο εν μέρη στο πρόβλημα της γεωργίας και των διεθνών αγορών. Δεν υπάρχουν μόνο οι διεθνής αγορά, δεν υπάρχει μόνο αυτό. Υπάρχει και η ευρωπαϊκή αγορά και η εθνική αγορά και πρέπει και η τοπική αγορά. Και με αυτές πρέπει να ασχοληθούμε και εκεί υπάρχει αστάθεια τιμών. Εσείς μιλάτε για αστάθεια τιμών μόνο στη διεθνή αγορά. Ε, θα πρέπει λοιπόν να έχουμε εργαλεία για να καταπολεμήσουμε την αστάθεια των ημών όχι μόνο στι διεθνεί αγορέ αλλά και στην τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή αγορά. Και όλα αυτά θα είναι αντικείμενο τη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε και των συμβαστικών λύσεων που πρέπει να βρούμε για το σύνολο των αγροτών και του κλάδου αυτού της οικονομίας. Έχετε κάποιες προτάσεις καταπολέμησης του φαινομένου αυτού και εδώ είναι η δεύτερη μου παρατηρήση. Και εδώ οι προτάσεις αυτές έχουν να κάνουν μόνο με την ιδιωτική σφαίρα. Η λύση για την αστάθεια των τιμών βρίσκεται και ε, στα μεικτά καθεστώτα και σε κατελάχιστον σε, στις διεθνείς σχέσεις των χωρών. Θα πρέπει να υπάρχουν και αυτά και όχι μόνο ο ιδιωτικός τομέας στην έκθεση. Βλέπετε τι γίνεται στον γαλακτοκομικό τομέα και πόσο έχει πληγεί από την κρίση. Βλέπετε τι γίνεται ε, στον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται διάφοροι ανταγωνιστές μας σε άλλες χώρες του κόσμου που μιλούν για μια δημόσια γεωργική πολιτική. Δεν πρέπει να περιοριστούμε ε, στον κλάδο της αγοράς μόνο και να μην μιλήσουμε καθόλου για τον δημόσιο φορέα για τη δημόσια πολιτική. Εγώ δεν είμαι κατά ε, της ρύθμισης από την αγορά. Υπάρχει και καλύτερη οργάνωση όμως των κλάδων. Σήμερα, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι αυτή η προσέγγιση της αγοράς, π.χ. στο γαλακτοκομικό τομέα, δεν αρκεί. Είναι σαφές αυτό είναι δύσκολο να επικαλωστούν το άρθρο 122 της κοινή οργάνωσης αγοράς στο γαλακτοκομικό τομέα. Δεν είναι συγκυριακός ο χαρακτήρας, είναι δομικός, διαρθρωτικός του προβλήματος. Ως προς το Ταμείο Ελληνοβοήθειας και τις ασφαλίσεις, να σας πω ότι κάνω την ίδια διαπίστωση. Η αγορά δεν λύνει τα προβλήματα από μόνη της. Και στην αμπελοϊνοκαλλιέργεια, πόσο μάλλον, υπάρχουν αγρότες που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά ε, τα εργαλεία. Το λέω για να εμπλουτίσω τη συζήτηση για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που είναι το θέμα της αστάθειας των τιμών. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Δυσκολεύτηκα να σας ε, διακόψω γιατί ήσασταν, ε, είχε, είχε πολύ ζωντάνια ο λόγος σας. Η κυρία Έρανθ Γκαρθία. Ευχαριστώ. Εγώ νομίζω ότι η απορρίθμιση της αγοράς είναι αυτή που καταφέρει τα πλήγματα τα, των οποίων γινόμαστε μάρτυρες. Αυτό που ζούμε από το 2003 ε, τώρα παίρνει σάρκα και οστά και γι' αυτό έχει έρθει και μας έχει πέσει το κεφάλι αν θέλετε. Ε, η κοινή γεωργική πολιτική θα χάσει εάν ε, πάει προς το Farm Bill των ε, Ηνωμένων Πολιτειών. Ίσως έχει έρθει η στιγμή να έχουμε συστήματα διαχείρισης κινδύνου και αυτό να είναι το μέλλον για την κοινή γεωργική πολιτική. Συμφωνώ με το θέμα των ασφαλίσεων. Όμως έχουμε π.χ. χώρες όπως η Ισπανία όπου τα συστήματα ασφάλισης λειτουργούν μια χαρά. Άρα, εάν πρόκειται κάτι να φτιάξετε στην Ευρώπη ή κάτι να φτιάξουμε, τουλάχιστον να συμβαδίζει και να συμφωνεί με χώρες όπου το σύστημα λειτουργεί καλά όπως η δική μας. Από εκεί και πέρα θα πρέπει οι αγρότες να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και όντως έχουν οργανώσεις ε, παραγωγών και πρέπει αυτές να τις ενισχύσουμε και να ενισχύσουμε και τις συμβασιακές σχέσεις, τη συμβασιοποίηση. Συμφωνώ με αυτές τις προτάσεις. Πρέπει να γίνουν βήματα σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας, όχι μόνο στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά μέχρι και τον τελευταίο κρίκο ε, της αλυσίδας, για να μην υπάρχουν κάποιοι που επιτίδη, που εκμεταλλεύονται ε, την αστάθεια των τιμών. Το παρατηρητήριο τιμών ε, γάλακτος είναι κάτι το πολύ θετικό και μπορούμε να το έχουμε και στους άλλους κλάδους της γεωργικής οικονομίας, όχι μόνο στο χείριο κρέας ή το ή άλλους κλάδους, αλλά και στα οποροκυπευτικά. Να έχουμε παρατηρητήρια τιμών και να έχουμε και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, έτσι ώστε να αντιδρούμε εγκαίρως. Να ε, χρησιμεύει δηλαδή αυτό το σύστημα παρατηρητηρίων των τιμών. Ε, όχι μόνο στηρίζω την πρόταση της κυρίας Δελαέ αλλά την εμπλουτίζω και με διάφορα άλλα στοιχεία που μπορεί να είναι θετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Τις γνωρίζουμε αυτές τις πληροφορίες σε γενικές γραμμές. Ωστόσο, η Επιτροπή, ξέρετε, πολύ συχνά ε, περιμένει το πρόβλημα να λυθεί από μόνο του, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Και η έγκαιρη παρέμβαση είναι λιγότερο δαπανηρή και περισσότερο αποτελεσματική. Πρέπει να δρούμε πιο γρήγορα. Ο κύριος Θεραμπέλα, παρακαλώ. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Δεν θέλω να τσακωθώ. Δεν είμαι Γάλλος, μιλώ γαλλικά, αλλά δεν θα μιλήσω για την γαλλική πολιτική. Όταν η κυρία Ντελαεμίλα αναφέρεται στους εμπειρογνώμες που ήρθαν στο κοινοβούλιο, είπε ο κύριος Σαλμά αναφέρεται, δεν θα λύσει αυτός ε, το θέμα της ε, σχετικότητας. Είναι, είναι υπερφελελεύθερος που λέει ε, ότι πάντα μπορεί να κάνει πολλοί πωλήσει ε, με προθεσμία. Αν αυτός είναι ο εξπέρ, τη βάψαμε. Ο κύριος Χανιώτης ε, ήρθε στην Επιτροπή Γεωργίας, ήταν διάφοροι συνάδελφοι, ο κύριος υποστήριξαν το, το TTIP που θα διαλύσει ακόμα περισσότερο τις τιμές. Το Farm Europe δεν ξέρω ποιοι είναι, είναι ε, πάντως δεν είναι υπερασπιστές της, ε, των γεωργών. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι αυτό. Είναι βεβαίως πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλίας, αλλά η μείωση της αστάθειας των τιμών σημαίνει έμεσα να δώσουμε ε, μία σταθερότητα στα εισοδήματα. Αυτό δεν συμβαίνει όμως γιατί η κυρία ε, Ντελαέ λέει δεν θα χτυπήσουμε τις χαμηλές τιμές. Τότε τι μήνυμα περνάμε στους γεωργούς. Τους λέμε ότι δεν θα κάνουμε τίποτα, κάνουμε μια, μια έκθεση που είναι κατά της αστάθειας αλλά λέμε χαμηλές τιμές. Συμβασιοποίηση. Ε, το σημείο 1 προφανώς είναι του κ. Σαλμά. Θεωρεί αναγκαίο ότι υπάρχει μια αστάθεια, μόνιμη αστάθεια στη γεωργία και αυτό είναι κανόνα. Ναι, μια κάποια, όχι πάντα. Ε, μετά, σημείο 2 διαπιστώνει ότι η Ενένωση συμβάλλει οικονομικά σημαντικά για να αντιμετωπιστεί η αστάθεια των τιμών. Αυτό είναι κάτι ωραίο, καλό για το αναφέρετε. Οργάνωση των ε, ε, τομέων και συμβασιοποίηση. Δεν αρκεί. Το δείχνουμε. Δεν αρκεί απλώς να προσπαθούμε να δώσουν βάρο στου γεωργού σε σχέση με άλλου φορεί Ποτέ θα έχουν το βάρο αν δεν παρέμβει ο δημόσιο, το δημόσιο. Δεν αναφέρεται το δημόσιο. Διαχείρι, εργαλεία διαχείριση κινδύνων. Ναι, ωραία, οι ασφάλειες, η ασφάλιση ένα κομμάτι τη λύση. είναι, δεν είναι η λύση. Περιοριστικό, αλλά μπορεί να το εξετάσουμε περαιτέρω. Παρατηρητήριο τιμών. Το παρατηρητήριο παρατηρεί. Άρα Ωραία είναι η παρατήρηση, αλλά δεν χρειάζεται την παρατηρούμε, ξέρουμε ποιε είναι οι τιμέ. Κυρία συνάδελφε, λοιπόν, ε, ελπίζω ότι χάρη στους συναδέλφους θα υπάρξει μια πλειοψηφία που θα επιτρέψει η έκθεση να είναι ένα έμβριο λύση. Το να διαπιστώνουμε ότι υπάρχει σοβαρή κρίση δεν μας νοιάζει, το ξέρουν οι γεωργοί. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συμβάλλουμε από κοινού για μια λύση και στη βάση αυτή η έκθεση που στηρίζεται, επαναλαμβάνω, σε εμπειρογνώμονες την ειλικρίνα των οποίων αμφισβητώ, ε, απέχει πολύ από αυτό που θα περιμένουμε και ελπίζω να το διορθώσουμε μέσω των τροπολογιών και των συμβιβασμών που θα προκύψουν. Ευχαριστώ. να προτείνω να συναντηθείτε και να συζητήσετε τα θέματα αυτά με ένα καφεδάκι. Προφανώς μπορείτε να εκφράσετε την άποψή σας. Ε, ε, δημοκρατία έχουμε. Κύριε Κιλέρα. Ε, Ευχαριστώ. Οι συνάδελφοι σχολίασαν την έκθεση αυτή ήδη. Έχει πολλά σημεία σύγκλησης με την έκθεση που συζητείται τώρα στην Ολομέλη και που μπορούμε να είμαστε γιατί είμαστε εδώ. Την ε, διαχείριση αξιών, την ε, αλυσίδα αξιών. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις. Συμφωνώ ωστόσο με τον συνάδελφο κύριο Ταραμπέλα ότι είναι χαμηλότεροι των προσδοκιών και των αναγκών. Η αστάθεια των τιμών ε, που λαμβάνουν οι γεωργείς ε, οφείλεται κατά βάση διότι έφυγαν όλοι οι μηχανισμοί του δημοσίου. Οι παρεμβάσεις ε, βρεθήκαμε δηλαδή στην έρμεα της αγοράς. Οι γεωργοί ενώπιον της καταστάσεως αυτής δεν πιστεύω ιδιαίτερα στην ιδιωτική ρυθμιστική πολιτική. Κώδικες καλής πρακτικής, ωραίοι είναι, αλλά δεν, δεν ε, επιτυγχάνουν στόχους. Αν θέλουμε λοιπόν να παρέμβουμε και να, έχουμε, να έχει σημασία η παρέμβασή μας, πρέπει να μπαίνουμε στους μηχανισμούς διαχείρισης αγοράς. Δεν θελήσαμε να το πειράξουμε στην τελευταία με, με, μεταρρυθμίση και είναι η βασική αδυναμία του κλάδου. Εξού και η αστάθεια των τιμών. Γιατί αυτό που λέμε είναι να οργανώνονται γιατί η αγορά είναι αγορά και όποιος δεν ε, αντιδρά πέφτει. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια μνήα στον τον ανταγωνισμό τρίτων χωρών γιατί και αυτό προκύπτει στην εσωτερική αγορά. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι η έκθεση μπορεί να κάνει ωραία συζήτηση για τη γεωργία στην Ευρώπη, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί και αυτό είναι που ζητούν οι γεωργοί. Η κατάσταση σε κάποιους κλάδους ιδίω είναι εξαιρετικά σοβαρή. Δεν αρκούν τα λόγια. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζουφίλα, ευχαριστώ. Νομίζω ότι η συζήτηση είναι και ζωντανή και πολύ ενδιαφέρουσα. Αποδεικνύει δε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια έκθεση που συνδέεται με την πραγματικότητα. Καταρχάς θεωρώ σημαντικό να υπογραμμίσουμε, το είπαν και προγενέστες συνάδελφοι, ότι η αστάθεια των τιμών έχει αποκτήσει διαθωτικό πλέον χαρακτήρα και είναι τόσο σοβαρή που πρέπει να αντιμετωπιστεί δεν αρκούν πλέον ε, μέτρα εφάπαξ για αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων. Μια, ένα τέτοιο δεν ε, λύνει την κατάσταση. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα σταθερό για προστασία των γεωργών μας. Μεταξύ άλλων και γιατί τα επίγοντα μέτρα φτάνουν με καθυστέρηση. Συχνά οι εκμεταλλεύσεις είναι κλειστές, ιδίω οι πιο μικρές. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προβλέψει ε, για το σκοπό αυτό μηχανισμούς απλοποιημένους. Εμείς μιλάμε για απλοποίηση πάντα. Συχνά ξεχνάμε να το θυμίσουμε στην Επιτροπή. Ε, η απλοποίηση είναι ένα όρος που πάντα να έχει υπόψη τη μοιρό κυρίω για τις ρήτες διαφυγή των συμφωνιών εμπορικών αλλαγών που πρέπει να είναι πιο ευέλικτε. Στην περασμένη περίοδο είδαμε πόσες ελλείψεις διαπιστώθηκαν που δεν μπορούσαν να καλυφθούν μέσω των ρήτων διαφυγής. Πρέπει να υπάρξει μια πολιτιστική αλλαγή επίσης, ενθαρρύνοντας ε, τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις να λειτουργούν με επιχειρηματικό τρόπο Εδώ σημαντικό ρόλο παίζουν οι νέοι που έρχονται στη γεωργία με νέο τρόπο, με πιο managerial τρόπο. Το θέμα της μεγάλης, των μεγάλων ε, αλυσίδων δια, διανομής είναι ένα σημαντικό θέμα. Κλείνω λέγοντας ότι πρέπει να δώσουμε πρόσβαση σε ευέλικτα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Η γεωργία πρέπει να είναι εξαιρετικά, η χρηματοδότηση γεωργίας πρέπει να είναι εξαιρετικά εύκαμπτη, αλλιώ θα έχουμε μπροστά μας μια κρίση που θα είναι μόνιμα διαθεωτική. Η κυρία Καστίνια, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πολλά υπόθηκαν ήδη θα ήθελα να ξαναευχαριστήσω την ε, συναδελφό μας την Οζελίκ Τελαή για την έκθεση αυτή. Πολλά από τα περιεχόμενα της έκθεσης ε, ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση και θα πρέπει να τα στηρίξουμε. Πολύ σύντομα βρίσκω σωστό να εξετάσουμε πιο προσεκτικά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να δούμε που υπάρχουν ρητές δυνατότητες ε, να πάρουμε πόρους από εδώ για την ε, γεωργία. Δεν αποκλείεται η γεωργία. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαθέτει χρήματα σε πολλούς τομείς. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε με τρόπο καινοτόμο. Γενικά πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι στην έκθεση αυτή. Όσον αφορά την εφαρμογή, αυτά που καταγράφει η Κομισιόν, ε, το τελικό αποτέλεσμα συχνά είναι απλά ένας μικρός συμβιβασμός. Νομίζω λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει με τόλμη να απαιτήσει ε, μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε ε, καινοτομίες, πώς μπορούμε να στηρίξουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις που μπορούν να ωφελήσουν τη γεωργία. Θα πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε τις γεωργικές νεοφυείς επιχειρήσεις ε, να τις συνδυάσουμε με νέους τομείς και να εντοπίσουμε εδώ τις ευκαιρίες. Νομίζω ότι σκεφτόμαστε πολύ συντηρητικά μερικές φορές ε, και ακολουθούμε τις παραδοσιακές οδούς και νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πιο προσεκτικά το θέμα των γεωργικών αγορών. Επίσης ε, θα πρέπει να στηρίξουμε τους νέους ε, και να δώσουμε εδώ μια νέα προοπτική. Αυτό θα πρέπει να είναι το κλειδί για την πολιτική μας στον τομέα αυτών στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε και Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, ε, θα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφα για τη δουλειά που έχει κάνει, αλλά δεν αρκούν αυτά που έχουμε. Ήδη έχουμε συζητήσει μία έκθεση για το γάλα και τον ανταγωνισμό και διαπιστώσαμε ότι δεν αρκούν τα χρήματα στον τομέα αυτών. Οι παραγωγοί έχουν διαφορετική θέση από τα μεγάλα γαλακτοκομεία τι νόημα έχουν όλα αυτά λοιπόν ε, τη στιγμή που ο ε, παραγωγός ε, γάλακτος αντιμετωπίζει έναν κολοσσό και δεν μπορεί να συνομιλήσει επίσης όρις. Όπως στη Δανία που υπάρχει μία μεγάλη γαλακτοκομία. Για μένα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, η έκθεση αυτή έχει προσανατολισμό την ε, συνένεση, λέμε ότι θέλουμε να προωθήσουμε ένα κλίμα διαλόγου, αλλά δεν αρκεί κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Ε, διακυβεύεται η ύπαρξη των ε, παραγωγών. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μέτρα. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, είναι πολύ ασθενής η διατύπωση στην έκθεση αυτή, λαμβανωμένης υπόψη της κατάστασης οι παραγωγοί θα πρέπει νομικά να έχουν διαφορετικό καθεστώς. Επίσης, ε, συζητάμε το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αλλά είναι όντως η σωστή κατεύθυνση το ότι καταργούμε όλο και περισσότερο την οργάνωση της αγοράς. Μήπως η απελευθέρωση και η κατάργηση της οργάνωσης της αγοράς ε, είναι λάθος δρόμος. Μήπως πρέπει να συζητήσουμε ποια κατεύθυνση θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και όσον αφορά τη διαχείριση του κινδύνου. Ναι, είναι πολύ ωραία όλα αυτά, το, τα ταμεία, η αμοιβαιότητα ακούγονται πολύ ωραία, αλλά πρέπει να περιγράψουμε πιο αναλυτικά τι ακριβώς εννοούμε. Ποιος ε, θα χρηματοδοτήσει τα ταμεία αυτά. Και Όσον αφορά την ασφάλιση στο σημείο 17, λέμε ότι δεν θέλουμε να χαθεί η δυναμική, αλλά δεν υποφέρουν και οι άλλοι από την αστάθεια των τιμών. Πού θα πρέπει να επενδύσουμε λοιπόν αυτό, είναι ένα συνολικό πρόβλημα στην αγορά. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να προσθέσουμε κάτι στη διατύπωση. Μπορεί κανείς να ε, ασφαλιστεί σε περίπτωση ε, χαλαζιού ή ε, καταστροφής παραγωγής, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε ασφάλιση κατά του Πούτιν. Θα πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε τις αγορές. Και επίσης η παρακολούθηση της αγοράς είναι ωραίο πράγμα. Η παραγωγοί μπορούν να το κάνουν αυτό όταν κοιτούν τον ισολογισμό τους. Ε, θα πρέπει όμως να έχουμε ένα εργαλείο της αγοράς ώστε να υπάρχει ένας μηχανισμός που να τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση προβλημάτων και όχι απλά να παρακολουθούμε. Νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσουμε δόντια στην έκθεση αυτή, να το πω έτσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Μπούντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά υπόθηκαν απόψε για το θέμα αυτό που συζητάμε από ε, την ε, αρχή που δημιουργήθηκε η Επιτροπή μας. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να καταπολεμήσουμε την αστάθεια των τιμών. Στη Ρουμανία υπάρχουν παραγωγοί που δεν μπορούσαν ούτε να πουλήσουν μια αγελάδα για 200 ε, ευρώ, που είναι μια ελάχιστη τιμή. Τι θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν, το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη αγορών για τη διάθεση των προϊόντων. Και δυστυχώς μερικές φορές είχαμε πιο πολύ πυροσβεστική αντιμετώπιση, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε μακροπρόθεσμα, ώστε να αποφύγουμε ή να μετριάσουμε κάποιες από τις κρίσεις που πιθανόν να εμφανιστούν και θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τους γεωργούς ώστε να μπορούν να δημιουργούν οργανώσεις παραγωγών. Έχω επισκεφτεί πολλές εκμεταλλεύσεις στο Βέλγιο και στη Γαλλία και έχω δει γεωργούς ε, που μπόρεσαν ε, να δημιουργήσουν τις δικές τους ε, εγκαταστάσεις μεταποίηση, ώστε να μην εξαρτώνται από κάποιον εξωτερικό παράγοντα που να κάνει την μεταποίηση. Θα πρέπει λοιπόν να κλείσουμε τον κύκλο εδώ στην παραγωγή μιλάμε για χαμηλές τιμές, αλλά τι είναι η χαμηλή τιμή σε σχέση με τι. Θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο κόστος του κάθε προϊόντος και την τιμή πώλησής του. Και τότε θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την αστάθεια στις τιμές. Ευχαριστώ. Η κυρία Μόη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι προφανές σε όλους και ιδίως στους γεωργούς ότι η αστάθεια των τιμών εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την συνέχιση της γεωργίας στην Ευρώπη. Η παγκοσμιοποίηση με πολιτικά μέτρα όπως το ρωσικό εμπάργκο και φυσικοί ε, κανόνες ε, δημιούργησαν ακόμα καλύτερη αβεβαιότητα στον τομέα. Και η Ευρώπη, ωστόσο, μέχρι τώρα λειτουργήσε με μειωπικό τρόπο. Η ΚΑΠΑ δεν έδωσε τις, ε, τους καρπούς. Στον, ε, ο κλάδος, ε, το γαλακτοκομικός κλάδος, στην ακρόαση πριν δύο εβδομάδες στις Βρυξέλλες, έκαναν προβλέψεις αποτελεσμάτων που θα εμφανιστούν μόνο το 2020 κατά την άποψή τους. Δεν μπορούμε όμως να περιμένουμε. Δεν μπορούν οι γεωργοί να περιμένουν. Αν θέλουμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο, η κρίση αυτή να μας ξεφύγει, θα πρέπει στο κέντρο της κοινή γεωργικής πολιτικής να βάλουμε τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την εγγύηση, των, με την ε, αστάθεια των τιμών, εξασφαλίζοντας ε, ομοιογενή μέτρα σε όλα τα κράτη-μέλη, δίνοντας μεγαλύτερη διαφάνεια στους γεωργούς και καταναλωτής με νέα και πιο ε, και πιο εύκολα μέτρα. Ιδίω ε, χρειάζεται σε κάποια κομμάτια της Ευρώπης ε, να ε, γίνονται με σοβαρότερο τρόπο οι έλεγχοι. Γιατί συχνά υπάρχουν απάτες από οργανωμένο έγκλημα, η μαφία για παράδειγμα. Η απάτη αυτή έχει υπεξαιρέσει τεράστια δημόσια κονδύλια από ανθρώπους ε, που τα χρειάζονται, τους γεωργούς. Και αυτό υπό, τα, υπό τους οφθαλμούς όλη της Ευρώπης, που δεν έκανε πολλά πράγματα τους ελέγχους μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τέσσε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε ενδιαφέρον τη συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ντελαέ για τις ε, προτάσεις της. Ε, μπορούμε να υποβάλουμε περαιτέρω προτάσεις και τροπολογίες, αλλά νομίζω ότι το κείμενο αυτό αποτελεί πολύ καλή βάση για τις εργασίες μας. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετείχε από την αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να παραμείνει, αλλά εγώ από μικρό παιδί βλέπω την ε, ε, εξέλιξη της ε, γεωργικής πολιτικής. Ε, έχουμε ένα εκατομμύριο Είχαμε ένα εκατομμύριο ε, αφιερωμένο γάλα ε, ή μπούτυρο ε, στις αποθήκες μας και γι' αυτό θα πρέπει να επιλέξουμε διαφορετική οδό. Και θα ήθελα να μιλήσω για την αλυσίδα της αγοράς. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Αυτά που άκουσα από τους παραγωγούς γάλακτος τις τελευταίες εβδομάδες είναι ανατριχιαστικά. Ένα παράδειγμα να σας δώσω. Πριν έξι εβδομάδες είχαν ένα προϊόν που στήχιζε 2 ευρώ 90 cents. Αυτή ήταν ήδη ε, πολύ χαμηλή τιμή. Έξι εβδομάδες μετά ε, η μεγάλη αυτή αλυσίδα σούπερ μάρκετ είπε ότι αν δεν κατεβάσετε τη τιμή από 2,90 σε 2,80 τότε δεν ε, θα απολούμε πια το προϊόν. Οι, αλυσίδες, οι μεγάλες αλυσίδες δηλαδή έχουν ε, τόση ισχύ που είναι αδύνατο να διαπραγματευτεί κανείς μαζί τους. Άλλο παράδειγμα. Στην Γερμανία είχαμε δύο παραγωγούς για ένα συγκεκριμένο είδος στήριου. Αυτό λειτουργούσε επί πολλά χρόνια καλά η τιμή ήταν καλή, ε, αλλά κατόπιν ήρθε τρίτος παραγωγός, ε, διάθεσε στην αγορά έναν τόνο τυριού ε, σε χαμηλότερη τιμή και έτσι κατέρευσαν οι τιμές του τυριού αυτού. Ε, δεν νομίζω ότι αρκεί να υπάρχουν οργανώσεις παραγωγών. Θα πρέπει να λάβουμε μέτρα για τον περιορισμό της ε, ισχύω αυτών των μεγάλων αλυσίδων για να συνεχίσει να υπάρχει η Ευρωπαϊκή Γεωργία. Και επίσης ε, χρειαζόμαστε νέα φορολογική πολιτική. Ε, πριν δύο χρόνια ε, είχαμε μια καλή συμφωνία, οι ε, φόροι να πληρωθούν μετά από δύο χρόνια, αλλά φέτος που πρέπει να πληρωθούν αυτοί οι φόροι ε, είναι και κακή χρονιά. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τις μικρές εγκαταστάσεις και θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες και στον γεωργικό κοινωνικό τομέα. Θα πρέπει συγκεκριμένο ποσοστό των ε, φόρων από τη γεωργία να διατίθεται ε, για τον τομέα αυτών. Θα πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε αυτό. Επιπλέον ε, υπάρχουν τεράστιες ανισότητες στα κράτη-μέλη. Ο κύριος Τόρφμαν στο Νότιο Τυρόλο στην Ιταλία ε, γιατί παίρνει 60 ευρώ και στη Λομαρδία 600 ευρώ. Αυτές οι ανισότητες ε, θα πρέπει να εξαλειφθούν και στην ε, Γαλλία συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Ε, κοντά στο Παρίσι που δεν είναι και οι πιο φτωχές εγκαταστάσεις λαμβάνουν πολύ περισσότερα από ότι σε πιο απόμακρες περιοχές. Και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, το best seller της Γερμανίας αυτή τη στιγμή ε, είναι ε, για vegans, για χορτοφάγους που δεν ε, τρώνε ούτε γάλα και αυγά. Αλλά εάν το κάνουν αυτό οι Γερμανοί, τότε δεν χρειαζόμαστε ούτε γαλακτοκομία ούτε κτηνοτρόφους. Και το 75% των γεωργικών περιοχών είναι βοσκότοποι, οπότε ε, δεν θα ε, διατίθεται πια για την παραγωγή. Ε, χόρτο θα καλλιεργούμε και μην σας πω και τι χόρτο. Πιστεύω ότι θα πρέπει όλα αυτά να συγκεντρωθούν μέσα σε ένα βιβλίο ενδεχομένω. Ο κύριος Φλάναγκαν. Ξέρετε, όταν έρχεται κανείς εδώ και ακούει για την κρίση στην Γεωργία και ακούει τα διάφορα επιχειρήματα και ε, προβληματίζεται, ε, επανέρχεται και ξανακούει τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Εν πάση περιπτώσει, ο προβληματισμός είναι πότε επιτέλους θα δράσουμε. Θα μπορούσα να σας πω ότι είπε ο προηγούμενος ομιλητής πριν τα πει, γιατί ήξερα την άποψή του ήδη. Πρέπει να κάνουμε κάτι για το μέγεθος των σούπερ μάρκετ. Καλό είναι να μιλάμε για την ενίσχυση των παραγωγών, για να έχουν την ίδια πυγμή, αλλά τελικά θέλουμε κάποιοι να έχουν τόσο μεγάλη πυγμή όπως τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Δύο χρόνια είμαι εδώ και τα λέμε ξανά και ξανά και ξανά επιτέλους πότε θα κάνουμε κάτι για το μέγεθος των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ που γίνονται τελικά τέρατα ε, που επιβάλλονται στους πάντες στην αγορά. Ιδαλλιώς θα ερχόμαστε εδώ και θα συναντιόμαστε και θα συνοδριάζουμε και θα ε, ακούμε όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Μπορούμε επιτέλους να δράσουμε ή υπάρχουν καλές ιδέες. Μας ακούει κανείς. Και σύν της άλλης. Και στη δική μου χώρα, αλλά και στις άλλες χώρες μου λένε ότι ένας αγρότης παίρνει π.χ. 40.000 ευρώ το χρόνο και το άτομο δίπλα του δεν παίρνει τίποτα. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, όπου υπάρχει βοήθεια για τον έναν και όχι για τον άλλον, αυτό είναι δραματικό. Η βοήθεια που υπάρχει, υπάρχει για να επιβεώσουν οι αγρότες. Αλλά τα έχουμε πει αυτά εκατομμύρια φορές. Εγώ δύο χρόνια είμαι εδώ, κάποιοι από εσάς είστε εδώ 15 χρόνια και σίγουρα ξέρετε πολύ καλά όλα τα επιχειρήματα. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Η ισορροπία είναι το πιο σημαντικό. Κύριος Γιάρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγώ ανήκω σε αυτούς που χαίρονται για την συζήτηση αυτή. Όπως είπε και η συγγήτρια, θα έχουμε μεγάλη συζήτηση. Σημείωσα και αυτά που είπε ο Άλπερτ Ντες. Άλλωστε και η κοινή οργάνωση της αγοράς ε, δεν ήταν ούτε και αυτή ο παράδεισος. Δεν λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Είχαμε σταθερές τιμές, ε, αλλά λίγο πριν την κατάργησή του είχε χρεοκοπήσει το σύστημα. υπάρχουν πολλές ανισορροπίες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, και τις οποίες δεν έχουμε αντιμετωπίσει με τα σωστά εργαλεία. Έτσι το περιγράφω ε, εγώ. Υπάρχει η ανισορροπία ανάμεσα στους παραγωγούς και τις μεγάλες ε, αλυσίδες. Αυτό συνδέεται με τον τρόπο σύναψης των συμβάσεων. η κοινή γεωργική πολιτική δεν είναι δίκαιη. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους μεγάλους και τους ε, μικρούς. Ε, όποτε δεν μπορούμε να εξηγήσουμε την κοινή γεωργική πολιτική λέμε ότι έχει εξελιχθεί στην ιστορία και έτσι έχει καταλήξει. Και θα πρέπει να τονίσουμε και την ευθύνη που φέρει ο ίδιος ο παραγωγός. Πάντως με ανησυχούν πολύ αυτά που περιέγραψε ο Αλπερτές. Έχουμε τεράστια ανισορροπία ανάμεσα στους παραγωγούς και την πυγμή που έχουν οι μεγάλες αλυσίδες. Εάν ε, δεν καταφέρουμε να αλλάξουμε την κατάσταση, τότε δεν θα έχουμε πια κοινή γεωργική πολιτική και δεν θα χρειάζεται καν να το συζητάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που δίνετε το λόγο στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούσαμε προσεκτικά και παρακολουθήσαμε προσεκτικά όλη αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε για την ενδιαφέρουσα έκθεση. Παρακολουθούμε στενά την έκθεση αυτή, γιατί το θέμα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ε, ειδικότερα στο πλαίσιο της ε, γεωργικής κρίσης και εκτιμούμε ιδιαίτερως το γεγονός ότι η έκθεση προσπαθεί να εστιάσει το ενδιαφέρον της ε, στα εργαλεία για τη διαχείριση της κρίσης και όχι μόνο στα κατεπήγοντα μέτρα και αυτό είναι καλό, θα δομήσει σωστά τη συζήτηση και θα μας βοηθήσει να έχουμε ένα σαφές ε, παραδοτέο από πλευράς της Επιτροπής σας. Όπως λέει λοιπόν η έκθεση, ήδη στην κοινή γεωργική πολιτική υπάρχουν εργαλεία τα οποία δυστυχώς δεν έχουν αξιοποιηθεί και ίσως μάλλον θα μπορούσαν να είχαν λύσει αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν ήταν και πολύ δημοφιλή. Και τέλος, για τη διαφάνεια. Δεν θα υποτιμούσα τον ρόλο της διαφάνειας. Η διαφάνεια δεν συνίσταται μόνο στην παρατήρηση του τι συμβαίνει, αλλά και στο μοίρασμα των πληροφοριών σε όλους τους παράγοντες. Υπάρχουν παράγοντες που δεν έχουν πρόσβαση σε όλη την πληροφορία. Και υπάρχουν παραδείγματα αποφάσεων που λαμβάνουν αγρότες στην Ευρώπη, χωρίς να είναι ενημερωμένοι για την ε, πραγματική κατάσταση της αγοράς από τους γαλακτοκομικούς και γαλακτοπαραγωγικούς συνεταιρισμούς τους, για παράδειγμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η διαφάνεια θα πρέπει να υπάρξει σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε παρατηρητήρια σε 17 κρατημέλη που λειτουργούν πολύ καλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο Λίαν συντόμως θα έχουμε παρατηρητήριο για το βόλιο και χείριο κρέας, ήδη το έχουμε για τα γαλακτοκόμικα και υπάρχει και το ε, άμις, το σύστημα πληροφοριών για τις γεωργικές αγορές κατόπιν της πρωτοβουλίας που εγκρίθηκε στο G20. Σας ευχαριστώ. Merci, Alors, je vais... Επόμενη ομιλήτρια, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, η συγγήτρια κυρία Ντελαέ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω συλλογικά και να μην ξεχάσω πολλά πράγματα γιατί πολλά έθιξαν οι προλαλήσαντες. Να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι αυτή η έκθεση δεν είναι έκθεση μεταρρύθμισης ή πλήρους ανανέωσης της κοινή γεωργικής πολιτικής. Στόχος της έκθεσης είναι να ασχοληθεί με το πρόβλημα της αστάθειας των τιμών. Τι θα πει αστάθεια, το εύρος διακύμασης που είναι πολύ μεγάλο και η συχνότητα με την οποία επανεμφανίζεται αυτό το φαινόμενο. Ε, αστάθεια δεν μιλούμε μόνο για τις πολύ χαμηλές τιμές αλλά και για τις πάρα πολύ υψηλές που και αυτό συμβαίνει. Βεβαίως αυτό το τεράστιο εύρος ε, καλύπτει ένα μέσο όρο τιμών που έχει πτωτική τάση και αυτό πράγματι είναι ανησυχητικό για τα εισοδήματα των αγροτών. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι εγώ είμαι αγρότης και έχω ζήσει διάφορες κρίσεις ε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παραμένει όμως η εκμετάλλευσή μου, παραμένει η επιχείρησή μου λειτουργεί παρά τις δυσκολίες και ο ιδιωτικό τομέας επιτρέπει να βρίσκουμε λύσεις. Δεν είναι αυτός σκοπός ο ιδιωτικό τομέας και δεν είναι το μοναδικό εργαλείο. Συμφωνώ με πολλούς από εσάς, είναι απαραίτητες αυτές οι προϋποθέσεις αλλά όχι επαρκείς και περιμένω τις τροπολογίες σας, τις προτάσεις σας έτσι ώστε οι απαραίτητες προϋποθέσεις να καταστούν και επαρκείς όχι μόνο αναγκαίες αλλά και επαρκείς για να βρούμε αρκετά εργαλεία. Πολλά εργαλεία της κοινής γεωργικής πολιτικής δεν τα έχουμε αξιοποιήσει και θα πρέπει να επιδείξουμε φαντασία και να προτείνουμε νέα εργαλεία. Το, η έκθεση που σας προτείνω είναι μια βάση συζήτησης έτσι ώστε να υποβάλλετε προτάσεις. Πολλής λόγος έγινε για την διαφάνεια και τη σχέση διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα. Δεν είναι αντικείμενο της έκθεσής μας. Ε, αντικείμενο της έκθεσης της κυρίας Μακίνες είναι αυτό. Και όταν είχα, ήμουν αρμόδια για γεωργικά θέματα σε εθνικό επίπεδο, είχα ασχοληθεί με αυτό το θέμα, αλλά δεν μπορούμε να το εξετάσουμε στην δική μου έκθεση. Θα πρέπει να βρεθεί όμως ένα νομοθετικό πλαίσιο. Συμφωνώ τους μαζί σας, δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Γεωργία ε, έρμεο στις αποφάσεις ενός μεγάλου ή λίγων μεγάλων ομίλων ε, διανομής. Η σχέση είναι πολύ άνηση και θα πρέπει ο νομοθετικός τομέας να παρέμβει ε, στο τομέα ε, ως προς αυτό. Συμφωνώ Κύριε Ταραμπέλα, είπατε ότι καλό είναι το να παρατηρούμε με τα παρατηρητήρια, αλλά όχι επαρκές. Αν ε, ε, δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν είμαστε σε θέση να πάρουμε αποφάσεις σωστές με βάση ε, την ιδιότητά μας ως παραγόντο της οικονομίας για να τοποθετηθούμε στρατηγικά στις αγορές. Η διαφάνεια είναι απαραίτητη και ε, σε κάθε στάδιο της θέσης σε εμπορία των προϊόντων. Ο Αλμπέχτο είχε πει, αλλά συμφωνώ με αυτή την ε, ιδέα, για τις οργανώσεις παραγωγών που δεν είναι επαρκή συνθήκη, είναι αναγκαία συνθήκη αλλά όχι επαρκής. Επομένως, Κάθε παράγον στην αγορά, όσο μικρός κι αν είναι, μπορεί να διαταράξει την αγορά γιατί δεν έχει ενημέρωση του τι κάνουν οι υπόλοιποι ε, παράγοντες στην ίδια αγορά. Όμως αυτό χρειάζεται εκβάθρον ανανέωση της κοινή γεωργικής πολιτικής και θα πρέπει να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα. Ενδεχομένως μακρηγορώ, ωστόσο οφείλω να πω ότι σε αυτή την έκθεση καλούμαστε να φανταστούμε εργαλεία διαχείρισης της αστάθειας των τιμών. Αυτό που σας προτείνω είναι ατελές, το γνωρίζω. Θα ήθελα όλοι να έρθετε στην ακρόαση και στο συνέδριο της 8ης Ιουνίου. Δεν μπορούμε να διώξουμε πυρογνώμονες, κύριε Ταραμπέλα. Εγώ είμαι υπέρ της πραγματικής θεώρησης. Η αγορά είναι έτσι όπως είναι, η οικονομία είναι παγκοσμιοποιημένη, μπορούμε να λυπούμαστε γι' αυτό όσο θέλουμε, αλλά πρέπει εκ των ενόντων να βρούμε λύσεις ε, επιδιόρθωσης αυτής της πραγματικότητας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, Θέλω να θυμηθείτε την ακρόαση στις 8 του μηνός. Να το θυμίσει παρακαλώ η γραμματεία σε όλους. Ε, λυπάμαι που δεν είχαμε τα της εκδηλώσει στο παρελθόν. Θα προσπαθήσω να είμαι παρόν. Εν γέννη, είναι καλό να ακούμε εμπειρογνώμονες και εταίρους μας, όπως τις είπα. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι οι οργανώσεις των γεωργών είναι σημαντικές, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε όλο το βάρος στις πλάτες μιας οργάνωσης παραγωγών είναι αδύναμη. Προθεσμία για τις τροπολογίες 13 του μηνός. Πρέπει να γίνει λίγη δουλειά βέβαια μετά την κατάθεση των τροπολογιών. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ την εισηγήτρια και για την έκθεση και τους συναδέλφους για την ε, συμμετοχή στη συζήτηση. Συνεχίστε την συνεργασία μέχρι τις 30 Ιουνίου. Στις 21 θα είναι η επόμενη συνάντηση της Επιτροπής μας, 20-21 Ιουνίου. Προχωρούμε στην συνάντηση των συντονιστών. Διακόπτουμε